Dear colleagues, we have to be... Στα αγγλικά η κυρία ε, Χάουκ, Και αγαπητοί συνάδελφοι, θα πρέπει να εφήσουμε ένα ισχυρό ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. The strongest ever, yes. Το στεναρότερο. Δεν ξέρω προηγουμένω τι λέγανε και ποιο. Εν πάση περιπτώσει, κάπω έτσι. Σαλβαδόρ γαρίγα. Λοιπόν, αγαπητοί συνάδελφοι, καλημέρα σας. Wir werden heute gemeinsam äh, durch diesen... Σήμερα θα διανύσουμε μαζί αυτή τη συνεδρίαση της Επιτροπής, διότι ο Πρόεδρος ήδη με μια αντιπροσωπεία έχει μεταβεί στη Σερβία και εργάζονται εκεί τόπου σήμερα και αύριο, οπότε κολλείται, δεν μπορεί να ε, βρίσκεται εδώ. Deshalb werden wir jetzt ähm, durch diesen Ausschuss gehen. Γι' αυτό λοιπόν θα διανύσουμε μαζί αυτό το διάστημα και μάλιστα πιστεύω ότι δεν θα εξαντλήσουμε και το χρόνο μας, εκτός ε, αν θέλετε να εξαντλήσετε όλα τα θέματα και έχετε και τρομερές νέες πτυχές να προσθέσετε από την περασμένη πέμπτη, που δεν το αποκλείω κιόλα. Ähm, να μην σας διαβάσω τώρα τις γλώσσες που έχουμε στη διάθεσή μας. Τα γνωρίζετε και μπορείτε να το διαβάσετε και στο Κόμπου News. Επίσης γνωρίζετε ότι μεταδίδονται όλες οι εργασίες μας στο διαδίκτυο. Επίσης δεν θα συνεδριάσουν οι συντονιστές μετά το τέλος της συνεδρίασης. Τουλάχιστον σε ό,τι αφορά τους συντονιστές τα γνωρίζουν οι ίδιοι. Τους τα έχουν διαβιβάσει οι συνεργάτες και οι βοηθοί τους. Και η επόμενη συνεδρίαση των συντονιστών θα γίνει στο Στρασβούργο τη Δευτέρα, την άλλη εβδομάδα. Äh, τα πρακτικά της περασμένης συνεδρίασης θα έχουν την μοίρα που τους επιφυλάσσουμε πάντα. Ε, όποιος δεν έχει καμία ένσταση αντίρρηση μέχρι το τέλος συνεδρίασης θα ε, θεωρηθούν τα πρακτικά εγκεκριμένα όσοι υπευλήθησαν. Έχετε λάβει όλο το σχέδιο ημερήσιας διάταξης και για πρώτη φορά, μια που έχουμε ορισμένους βουλευτές παρόντες, να αρχίσουμε με τις ψηφοφορίες για αλλαγή. Αρχίζουμε από τις ψηφοφορίες λοιπόν. Είναι το σημείο 9 στην ημερήσια διάταξη. Συγκρότηση του Ευρωπαϊκού Σώματος Εθελοντών Ανθρωπιστικής Βοήθειας. Η συγκήτρια είναι η κυρία Μαρία Μονίθ, καλύτερα συντάκτη αγνωμοδότησης, γιατί εμείς γνωμοδοτούμε. Έχετε όλοι τις κάρτες σας. Στα μηχανήματα άλλοι δεν έχουν καθόλου κάρτα. Καλά. Δεν είμαστε υποχρεωμένοι να ψηφίζουμε ηλεκτρονικά σε καμία ψηφοφορία εκτός από την τελευταία. Η τελευταία κάθε φορά ψηφοφορία πρέπει να γίνεται ηλεκτρονικά και της νομοδότησης και της έκθεσης. Όποιοι έχουν κάρτες παρακαλώ να τις βάλουν στη σχετική σχισμή και στα μηχανήματα και όσοι δεν έχουν κάρτα να φροντίσουν να ε, μετρηθούν και να στοιχηθούν με την εκάστοτε παράταξη. <laughs> Γεια! Για! Sorry? Ja. <laughs> Ε, Edith Herzog. Ja, Ja, gut. Okay. Nichtsdestotrotz, wir Είμαστε έτοιμοι. Αρχίζουμε λοιπόν. Παρά όλα αυτά και τις ε, απουσίες. Ε, παράγραφος 1. Η τροπολογία 1. Ψήφι υπέρ. Κατά. Αποχές. Ε, εγκριάζει Τροπολογία παριθμό 2. Υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Η τροπολογία υπερθμό 3 κατά αποχές εγκρίνεται. Η τροπολογία Α, μάλλον έχουμε τη νέα παράγραφο 1D με μια προφορική τροπολογία την οποία έχετε και γραπτά Είπε κατά αποχές εγκρίνεται. Και τώρα ερχόμαστε στον κανονισμό τροπολογία υπερφών 6 κατά αποχές εγκρίνεται. Antrag 7. Wer ist dafür? Η τροπολογία 7 υπέρ. Κατά. Αποχέ. Ε, εγκρίνεται. Η τροπολογία υπέρ 8 και 9 μαζί. Μπορούμε. Όχι. 8. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Τώρα η 9 υπέρ. Wer ist dagegen? Κατά. απόχέ. Εγκρίνεται. Η τροπολογία υπαριθμών 10. Με την ε, σχετική προφορική υπέρ. Κατά. Αποχε. Εγκρίνεται. Η τροπολογία υπαριθμών 11. Και πάλι με μια προσθήκη προφορική υπέρ. Κατά. άποχε εγκρίνεται. Η τροπολογία υπαριθμών 12 υπέρ. Κατά εποχές εγκρίνεται. Η τροπολογία 36 υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. 13 και 14 μπορούμε να τις ψηφίσουμε ομού. Ωραία, 13 και 14 υπέρ κατά αποχές δεν Η τροπολογία υπερθμών 15 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Η επόμενη έχει αποσυρθεί. Η τροπολογία υπερθμών 16 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται η τροπολογία του 17 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται η τροπολογία υπέρ 18 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται η τροπολογία υπέρ 38 μπορεί να ψηφιστεί ως προσθήκη ε, για τη 18 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Τώρα, έχουμε τις αιτιολογικές σκέψεις, ε, recitals. Ο κύριος Χάρτον έχει καταθέσει 16 παρακαλώ τροπολογίες. Μπορώ να τις θέσω όλες μαζί, αν σε ψηφοφορία. Ποιος είναι υπέρ των τροπολογιών του κυρίου Χάρτονγκ κατά αποχές. Ωραία, συλλήφθεν λοιπόν απορρίπτονται. Και ερχόμαστε στην τροπολογία υπαριθμών 4, ψήφι Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Η τροπολογία υπαριθμών 5, υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. Ή 35 τώρα, του κυρίου Κοσλόφσκι, υπέρ. Κατά. Αποχές. Και αυτή εγκρίνεται. Και τώρα, η 35 τωρα Το κύριο κοσλοφσκι υπερ παρακαλώ ψηφοφορία, όσοι έχετε κάρτες. Wir zählen θα σα μετρήσουμε λοιπόν όσο δεν έχετε κάρτα. Mhm. Ψηφίσαμε όλοι. Πέρας. 25 συν 4 υπέρ, μία ψήφος κατά και δύο εποχές. Δηλαδή 29 υπέρ, ένας ε, κατά και δύο εποχές. Kommen Λοιπόν, προχωρούμε. Τι έχουμε τώρα. Σύσταση προς την Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Εξωτερικής Δράσης σχετικά με την αναθεώρηση της οργάνωσης και λειτουργίας της. Η συγγήτρια είναι η κυρία Νέινσκι, απούσα. Δεν πειράζει όμως, θα ψηφίσουμε. Η τροπολογία 1. Υπέρ. Κατά. Τώρα αρχίζει το μέτρημα, αλλά χρειάζεται και παλήθευση. Η ηλεκτρονική που αρχίζει τώρα. τι ψηφίζουμε την τροπολογία υπαριθμών 1, στην παράγραφο 1. Όλα 1 είναι. Πρώτη παράγραφος, πρώτη τροπολογία. Λοιπόν, ψηφίσατε όλοι, ξέρουμε και ποιοι είναι οι τέσσερι χωρί κάρτα. Συντόνια, Μοργάντη, Ράιμερ, Μπέγκε και άλλο 16, 17 υπέρ και 14 κατά εγκρίνεται. Adopted δηλαδή. Τώρα έχουμε την τροπολογία υπαριθμών 2. Είναι συμβατή με την προηγούμενη. Μάλιστα. Ψηφίζουμε τη 2. Υπέρ. Κατά. Μάλιστα. Απλό ήταν αυτό. Αποχές. Απορρίπτεται. Η συμβαστική α. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Και ερχόμαστε μέσα στην παράγραφο 3 και συμβαστική β υπέρ. Κατά. Αποχ... Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Παράγραφος 3. Η τροπολογία υπέρ 10. Με μια προφορική τροπολογία. Υπέρ. κατά άποχες εγκρίνεται τροπολογία παριθμών 11 Επέ. πάλι με την προφορική που έχει εδώ κατά άποχες εγκρίνεται Η τροπολογία παρελθόν 12. Στην παράγραφο 4. ψήφιο Κατά. Αποχές. Απορρίψτε. Η τροπολογία παρελθόν 13. Πε. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Τροπολογία 14 σε δύο τμήματα. Τμήμα πρώτον υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. Το δεύτερο τμήμα υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. η τροπολογία περισσότερων 15. Το πρώτο τμήμα καλά υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Το δεύτερο τμήμα. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. Η τροπολογία 16 υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Η τροπολογία 17 υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Και τώρα η τελική ψηφοφορία. Ηλεκτρονικά παρακαλώ με κάρτες. Αρχίζει η ψηφοφορία. πέρασε 28 συν 4, 32 υπέρ. Μία ψήφος κατά και μία αποχή. Μάλιστα. Λοιπόν, πάμε τώρα για ψάρι. Δεν είναι εύκολα τα πράγματα με τα ψάρια συνήθως. Αλληλευτική συμφωνία με Μαδαγασκάρι. Την έχουμε ξανασυζητήσει την τελευταία φορά και είπαμε ότι ε, θέλαμε να αναβάλουμε την ψηφοφορία μας. Για να ζητήσουμε από την Επιτροπή Αλίας Αναβολή, όχι καταψήφιση. Να αναβάλουν και αυτή την ψηφοφορία. Γι' αυτό ε, θα ήθελα να σας προτείνω το εξής προς ψήφιση. να σας διαβάσω κάτι. Η Επιτροπή Προϋπολογισμών καλεί την Επιτροπή Αλίας ως καθήλυνα αρμόδια να προτείνει ε, το Κοινοβούλιο να αναβάλει την ε, συνένεσή του μέχρι να λάβουν χώρα δημοκρατικές εκλογές στη Μαδαγασκάρη και να αποκατασταθεί η δημοκρατική τάξη και πάλι. Δηλαδή αναβάλουμε την απόφασή μας μέχρι να επανέλθει η δημοκρατία στη χώρα, μέχρι τις εκλογές. Και βέβαια και υπό το φως των εξελίξεων και την έκβαση των εκλογών. Αυτό θα πρέπει να ψηφίσουμε. Συμφωνείτε, διαφωνείτε. Ποιος είναι υπέρ. Ο κύριος Χάρτον ζητάει το λόγο για διαδικαστικό. Χωρίς μικρόφωνο δυστυχώς. Πρόεδρε, θέλω να δω την πρόταση αυτή γραπτός πριν ψηφίσω, γιατί αυτά μας τα διαβάζετε ωραία, αλλά είναι προφορικά. können... Θα προσπαθήσω. Αν θέλετε μπορείτε να το αναβάλουμε και μέχρι το τέλος της συνεδρίασης που θα έχετε και το κείμενο γραπτός αλλά μπορώ αν θέλετε και πάλι πάρα πολύ αργά να σας αναγνώσω για να μπορεί ο καθένας να τα ακούσει στη μητρική του γλώσσα εάν συμφωνείτε και μετά γνωρίζετε τι ψηφίζετε. Η Επιτροπή Προϋπολογισμών καλεί την Επιτροπή Αλίας, που είναι επί της ουσίας αρμόδια, να προτείνει να βάλει το Κοινοβούλιο να δώσει συνένεση μέχρι ε, σότου διεξαχθούν δημοκρατικές εκλογές στη Μαδαγασκάρη και αποκατασταθεί η δημοκρατική τάξη. Κύριε Χάρτον, σας αρκεί αυτό ως επανάληψη. Είναι πολύ καλή η διερμηνία και καλά κάνετε και το ε, διαβάζετε, αλλά θέλω η επίσημη πρόταση να είναι και ένα επίσημο κείμενο για να ξέρω τι ψηφίζω και να κανονίσω την πορεία μου. Und ναι. Μα, αν συμφωνήσετε, ε, στα πρακτικά θα εγγραφεί το επίσημο κείμενο. Ποιος είναι υπέρ, λοιπόν, αυτό που σας ε, ανέγνωσα, ε, για να βολεί χωρί συνένεση. Κατά της πρότασης αυτή που σας διάβασα. Αποχές. Εγκρίνεται. Das. Ja, ja. I understood, I understood you. Ναι, ναι, κατάλαβα. Είστε κατά των δημοκρατικών δομών. Ναι, το πιες. Πάνω κάτω, αυτό θέλει το ΕΛΚ. Εντάξει. Πάμε τώρα στην επόμενη ψηφοφορία. Πάλι για ψάρια πρόκειται και πάλι για αλληλευτική συμφωνία. Ε, δεν είναι εταιρική συμφωνία, δεν αρνούμε να την χαρακτηρίσω εταιρική την αλληλευτική συμφωνία. Τώρα πρόκειται εδώ για τη Μαυριτανία. Δύο-τρεις ψηφοφορίες πρέπει να κάνουμε. Η πρώτη είναι για την τελευταία παράγραφο που έχουμε μια τροπολογία υπαριθμών 1 του κυρίου Τζοβάνι Λαβία υπέρ της ε, τροπολογίας αυτής. Ψήφι. Α, ηλεκτρονικά, ηλεκτρονικά. Σας παρακαλώ. Ο Μπέγκε δεν ψηφίζει. Με κάρτα χωρίς κάρτα. Χαίρεται κιόλας που έχει ξεχάσει την κάρτα του. Λοιπόν. Mm. Δεν χρειάζεται να μετρήσουμε ούτε τίποτα, γιατί είναι σαφές το αποτέλεσμα. Απορρίψετε. Ε. Τότε, τι θα ψηφίσουμε το σύνολο της νομοδότησης ή του πρωτοκόλου υπέρ. Κατά. Άποχες. Εγκρίνεται. Και τώρα η τελική ψηφοφορία. Ηλεκτρονικά. Παρακαλώ. Στο βαθμό του πρωτοκόλλου υπερ κατα αποχες εγκρινεται και τωρα η τελικη ψηφοφορια ηλεκτρονικα παρακαλω στο βαθμο του δυνατου Λοιπόν, αποτέλεσμα 23 υπέρ, 11 κατά, μία αποχή. Αυτό είναι το αποτέλεσμα. Εγκρίθηκε λοιπόν και αυτό. Και έχουμε τελειώσει έτσι την ώρα των ψηφοφοριών. Όχι. Τι άλλη ψηφοφορία έχουμε. Ε, sorry. Ah. Μόνικα, lass mal bitte Giovanni eben Έχουμε μια μεταφορά, Μόνικα, μια στιγμή ε, το Τζοβάνι, γιατί έχουμε μεταφορά αίτηση Μια μεταφορά. Είναι η μεταφορά υπαριθμών 1 κάθετος 2013. Και θα μας πει ο εισηγητής αν θα πρέπει να ε, την υπερψηφίσουμε ή να την απορρίψουμε. Lo storno è relativo al trasferimento di... Ναι, λοιπόν, πρόκειται για μεταφορά απορών υπέρ των άμεσων πληρωμών προς τους ε, γεωργούς, δηλαδή πρώτος πυλώνας. Πρόκειται για πόρους που προέρχονται από τη Συμφωνία Αναδιάρθρωσης ε, του τομέα της ε, ζάχαρης στην Ευρώπη που προέβλεπε στο συμπέρασμα, στο τέλος δηλαδή του 2012 και οι πόροι έπειτα μεταφέρθηκαν στον προπολογισμό του 2013. Προβλεπόταν οι επιπλέον αυτοί οι πόροι, αν μάλλον υπήρχαν υπόλοιπα, αυτά θα χρησιμοποιούνταν από τον Ευρωπαϊκό Προπολογισμό και σε αυτή την περίπτωση ζητείται η μεταφορά υπέρ του καθεστώτος άμεσων πληρωμών που ήδη είχε υπάρξει τέτοιο αίτηση μεταφοράς. Από πλευρά μου δεν υπάρχει καμία δυσκολία, λοιπόν μπορούμε να το εγκρίνουμε. Wenn wir unserem folgen, αν θέλουμε να παρακολουθήσουμε τον εισηγητή μας και να ακολουθήσουμε αυτό που μας λέει, ψηφίζουμε λοιπόν υπέρ. κατά άποχες με μία ψήφο κατά εγκρίνεται όπως προτάθηκε. Τώρα όμως τέλειωσαν πραγματικά οι ψηφοφορίες, έτσι δεν είναι. Και συνεχίζουμε στην κανονική ημερήσια διάταξη. Το σημείο υπαριθμών 7. Γνωμοδότηση είναι και αυτή με θέμα... Α, σε ποια επιτροπή γνωμοδοτούμε, υποθέτω στην Επιτροπή Απασχόλησης. Ε, συντάξεις γνωμοδότησης είναι ο Ντέρεκ Βον. Το θέμα είναι το Ταμείο Ενίσχυσης των Απόρων στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Παρακαλώ, ο Ντέρεκ. Okay, uh, thank you, Chair. As... Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Όπως είπατε σωστά, πρόκειται για μια σύντομη γνωμοδότηση για την Επιτροπή Απασχόλησης και προσπάθησα να καλύψω κάποια ευρεία θέματα. Ε, προφανώς αυτά, σχετίζονται, ε, αυτά που σχετίζονται με το θέμα του προπολογισμού. Καλωσορίζουμε τη δημιουργία αυτού του ταμείου που αντικαθιστά το προηγούμενο πρόγραμμα επιστημιστικής βοήθειας και επίσης καλωσορίζουμε την διεύρυνση του πεδίου του προγράμματος ώστε να καλύπτει όχι μόνο επιστημιστική βοήθεια αλλά και τους άστεγους αλλά και την ηλική στέρηση των παιδιών. Θα γνωρίζουν οι συνάδελφοι ότι στην διάσκεψη κορυφής και 8 η Φεβρουαρίου το Συμβούλιο στήριξε τη συνέχιση του προγράμματος αυτού αλλά είπε ε, ότι θα πρέπει στο μέλλον να χρηματοδοτηθεί από το, ταμείο, ε, το Κοινωνικό Ταμείο. και ότι τα χρήματα αυτά θα, έμεναν, θα, θα ήταν συγκεκριμένα. Όσον αφορά την μείωση του συνολικού ποσού στα 2,5 ε, εκατομμύρια, σημαίνει πως αυτή τη στιγμή σημαίνει πως θα κατέβουμε στα 3 1,55 εκατομμύρια ευρώ ετησίως. Ορισμένοι συνάδελφοι θα προτιμούσαν να μείνουμε στο ποσό του, των 3,5 δις για να συνεχίσουμε την εμφιστάμενη χρηματοδότηση. Επίσης, στη γνωμοδότησή μου αναφέρω κάποιες ανησυχίες όσον αφορά το διοικητικό φόρτο που σημαίνουν ε, ίσως οι νέες προτάσεις. Επειδή χρηματοδοτείται από το Κοινωνικό Ταμείο, πρέπει να είμαστε απόλυτα βέβαιοι ότι δεν θα υπάρχουν ε, πολλά εμπόδια και γραφειοκρατικός φόρτος ε, ε, προς τις ΜΚΟ ή τις φιλανθρωπικές οργανώσεις που θέλουν να ωφεληθούν από το συγκεκριμένο ταμείο. Επίσης, τα στόκ παρέμβαση θα πρέπει να χρησιμοποιηθούν από το πρόγραμμα αυτό δωρεάν. Δηλαδή, δεν θα πρέπει να θεωρηθούν ως επιβάρυνση για το πρόγραμμα μάλλον να θεωρηθούν ως προσθήκη στο πρόγραμμα και μην, να μην φεύγουν από συγκεκριμένους προπολογισμού των κρατών μελών. Στην τροπολογία 9 επίσης λέμε ότι οποιαδήποτε χρησιμοποιείται πόσα από το πρόγραμμα θα πρέπει να κρατηθούν και να δοθούν στα κράτη-μέλη που δεν χρησιμοποίησαν το κομμάτι τους, γιατί ορισμένα κράτη μπορεί να μην θελήσουν να το χρησιμοποιήσουν και αντί να χαθούν τα χρήματα ή να επανέλθουν στο κεντρικό ταμείο, να μπορέσουν να χρησιμοποιηθούν από άλλα που μπορεί να, χρη... να θελήσουν να χρησιμοποιήσουν παραπάνω χρήματα. Ένα σχετικά επίμαχο θέμα είναι αυτό που αφορά την συγχρηματοδότηση. Οι προτάσει τη Κομισιόν πρότειναν 85% των κονδυλίων θα πρέπει να προέρχονται από τα κράτη-μέλη και τα κράτη-μέλη να δίνουν το 15% των κονδυλίων. Ξέρω ότι η Επιτροπή Απασχόληση θα κάνει μια συζήτηση από αυτού και στι δικέ μου τροπολογίε, οι συνάδελφοι θα δουν ότι έχω διαγράψει τι αναφορέ στην συγχρηματοδότηση για αυτό το στάδιο. Θα γίνουν περαιτέρω συζητήσει και θα συνεχιστούν και διαπραγματεύσει με την Κομισιόν και το Συμβούλιο για το συγκεκριμένο θέμα. Η προθεσμία για υποβολή τροπολογιών είναι κιόλα αύριο, είναι κάπως στενά τα όρια, γι' αυτό και θα καλωσορίσω τα σχόλιά σας για τη γνωμοδότησή μου σήμερα, καθώς και τις τροπολογίες που μπορεί να υποβάλλετε πριν την αυριανή προθεσμία. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ. Έχει κανείς να πει τίποτα. Τζοβάνι, Λαβία. Und Jan Kozlowski. Sorry, first uh, Jan Kozlowski. Συγγνώμη, πρώτα ο Κοσλόφσκι και μετά Τζοβάνι Λαβία. Το Μινικρικέ και οι υπόλοιποι. Okay, uh, we will write it down. Uh, yeah, wir schreiben es auf. Ναι, ναι είστε πολύ, θα σημειώσουμε το όνομα του. Ε, Ευχαριστώ πολύ κυρία Πρόεδρε. Όπως και ο συγκητής έτσι πιστεύω ότι εντάσσεται στη στρατηγική του 2020 η χορήγηση πόρων του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου για τους πλέον απόρους. Σίγουρα θα πρέπει να πλουστεύσουμε στο δυνατόν περισσότερο το σύστημα. Το σύστημα όσο έχει αυτή τη στιγμή είναι άκρος πολύπλοκο και σε ό,τι αφορά τη κατανομή των κονδυλίων. Ε, μιλάμε για 2,5 δις για 7 χρόνια αλλά για όλα τα κράτη-μέλη. Αλλά και σε ό,τι αφορά το εύρος και το είδος ε, της ε, παρεχόμενης υποστήριξης. Θεωρώ λοιπόν, δεδομένης και της, ε, δεδομένης φύσης του Ταμείου, ότι η αύξηση των πιστώσεων πληρωμών θα ήταν θετική κατά 100% ε, των ε, αποδεδόμενων κονδύλων. Σε ό,τι αφορά σε ό,τι αφορά την αυτόματη διαδικασία, δεν θα ε, θεωρούσα σκόπιμο να εφαρμόζεται εδώ, διότι παρέχονται διαφορετικά υποστήριξη από αυτό το ταμείο. Αντιθέτω, ε, με το ταμείο συνεχίζει τα πράγματα διαφορετικά. Επίσης, Νομίζω ότι οι πληρωμές που αναφέρονται στο άρθρο 42 θα πρέπει να υποκίνονται σε μια προθεσμία 30 ημέρων. Επίσης, όλο το πλωμένο ανησυχεί είναι οι δείκτες. Οι για τα κράτη-μέλη. Πρέπει να περιληφθεί ως κριτήριο κατά την άποψή μου και η σχετική ένδυα, relative poverty. Τέλος, θέλω να στηρίξω τον κύριο Βον ως προς το πρόταση να μην βάλουμε υπερβολικού όρου εν καιρό κρίση, γιατί μπορεί να στερήσουμε ανθρώπου από του πόρου που έχουν ανάγκη. Ο Τζιοβάνι. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Όπω θα θυμούνται οι συνάδελφοι, αυτό το πρόγραμμα βοήθεια στου άπορου είναι ένα πρόγραμμα που κατά τη διάρκεια της, του προηγούμενη περίοδου προγραμματισμού ε, ε, ε, εντασσόταν στην γεωργική πολιτική και χρησιμεύε ώστε να χρησιμοποιηθούν αποτελεσματικά τα προϊόντα που αποσύρονταν από την αγορά και κατά και που με αυτόν τον τρόπο ετίθεντο στην διάθεση των απόρων μέσω δομών που διαχειρίζονται την επιστική βοήθεια. Τώρα το πρόγραμμα αλλάζει φύση και στην επιστηστική βοήθεια προστίθεται διάφορες άλλες δραστηριότητες. Γίνεται ένα κοινωνικό πρόγραμμα βοήθειας. Από τη μια πλευρά έχουμε λοιπόν διεύρυνση της γάμας των δραστηριοτήτων, από την άλλη έχουμε περιορισμό όμως των πόρων. Διότι όπως θα θυμάστε είχαμε ε, χρησιμοποιήσει στην προηγούμενη προγραμματική περίοδο 2007-2013 είχαμε 500 ευρώ, ε, εκατομμύρια ευρώ το χρόνο, ενώ ε, τώρα και στην τελευταία συμφωνία έχουμε 2,5 δις για το σύνολο της περίοδου. Χάνουμε δηλαδή 30%. Με λιγότερο 30% πόρους πρέπει να κάνουμε περισσότερα πράγματα. Όχι μόνο επισητιστική βοήθεια, αλλά και ένα πραγματικό πρόγραμμα κοινωνικής βοήθειας. Από την άλλη πλευρά θέλουμε ακριβώς να αυξήσουμε το επίπεδο χρηματοδότησης συγχρηματοδότησης γιατί αυτό σε ορισμένες περιπτώσεις αποτέλεσε εμπόδιο στην εφαρμογή του προγράμματος. Όλα αυτά είναι πράγματα δίκαια αλλά υπάρχουν κάποιες αντιφάσεις ανάμεσα σε όλα αυτά και γι' αυτό κατά τη γνώμη μου θα έπρεπε να δώσουμε μεγαλύτερη έμφαση στο πρόγραμμα σε αυτές που είναι οι πιο ουσιαστικέ πτυχές. Δηλαδή θα έδινα μεγαλύτερη προσοχή στην ε, επισητιστική βοήθεια, στη στήριξη δηλαδή των πρωταρχικών ε, αναγκών του πληθυσμού και γι' αυτό θα ε, ήθελα να εισάγω κάποια διόρθωση εδώ. Και έπειτα συμφωνώ στα όσα είπε ο Ντέρεκ για το θε... τα ποσοστά συγχρηματοδότησης, ότι δηλαδή θα ήταν σκόπιμο να ακολουθηθεί αυτή η κατένθεση σε σχέση με το θέμα των επιπλέον πόρων, που μάλλον που συνολικά διατίθεται για αυτό το πρόγραμμα, θα πρέπει να λάβουμε υπόψη ότι διανύουμε κρίση. Ο αριθμός των απόρων σε κοινοτικό επίπεδο, χρόνο με το χρόνο και κυρίως τα τελευταία χρόνια, αυξάνεται εντόνως και εμείς θέλουμε δηλαδή να κάνουμε περισσότερα πράγματα με λιγότερους πόρους σε μια περίοδο κρίσης. Κάτι νομίζω πρέπει εδώ να προσαρμόσουμε και να αναδιαρθρώσουμε και νομίζω πως θα πρέπει προς αυτή την κατεύθυνση να κινηθούμε. Ευχαριστώ. Ναι, ευχαριστώ πολύ. Ιζαμπέλ Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Θέλω να ευχαριστήσω τον εισηγητή για το σχέδιο έκθεσης που μας παρουσίασε. Συμφωνώ απόλυτα και σας ευχαριστώ κύριε Σικητά γιατί πρώτα απ' όλα επιλέξετε να είστε απλός και έχετε δίκιο γιατί πρέπει το κείμενο να είναι στο τέτοιο πιο απλό. Δεύτερον, συμφωνώ μαζί σας ε, προς τον κίνδυνο όπως είπε ο κύριος Λαβία πριν από μένα για τον κίνδυνο της συγχρηματοδότησης. Οι χώρες δηλαδή που έχουν ήδη οικονομικές δυσκολίες ε, θα είναι εκτεθειμένες σε ακόμα μεγαλύτερες. Και σίγουρα λόγω ακριβώ αυτή τη δύσκολη κατάσταση ε, θα έχουν ε, κοινωνικέ υπηρεσίε των χωρών αυτών δυσκολίε να ενισχύσουν του απόρου. Άρα τελικά τιμωρούμε ακόμη περισσότερο, κάνουμε ακόμη πιο δύσκολη την κατάσταση των ανθρώπων αυτών σε αυτέ τι χώρε. Ό,τι αφορά τα ποσά, επίση συμφωνώ με τι προτάσει Νομίζω ότι η πρόταση αυτή ε, είναι φιλόδοξη και δημοσιονομική ό,τι αφορά το δημοσιονομικό σκέλος. Ε, κάποιες απλουστεύσεις ε, καλό θα ήταν, αλλά συμφωνώ με το περιεχόμενο της έκθεσης, ιδίω για την γνωμοδότηση της Επιτροπής Προβλησμού που είναι τεχνικού χαρακτήρα μεν, αλλά αφορά μια πτυχή που έχει να κάνει με τη βοήθεια των θυμάτων της λιτότητας, γιατί ε, περί αυτού πρόκειται τελικά, δηλαδή όλο και περισσότεροι Ευρωπαίοι είναι θύματα της δημοσιονομικής αυστηρότητας, της δημοσιονομικής λιτότητας που επιβάλλει η Ευρώπη. Θα ήταν παράδοξο του προπολογισμού να λέμε ότι όχι. Είμαστε ήδη συνυπεύθυνοι και όχι μόνο αυτό, βάζουμε και οικονομικά όρια για να βοηθήσουμε ακόμα λιγότερο τα θύματα της ε, λιτότητας, για την οποία ευθυνόμαστε και εμείς σε έναν βαθμό. Αυτό το μήνυμα σε καμία περίπτωση δεν θα περνούσε ούτε από πολιτική, ούτε από κοινωνική πλευράς. Πολύ σωστά λοιπόν ε, τα λέει η και δεν θα καταθέσω καμία τροπολογία. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ πολύ. Τώρα ο Ντομινίκ Ρίκε, παρακαλώ. Σας ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε. Θέλω να ευχαριστήσω τον Τέρικ Βον για την έκθεσή του που να βρίσκει σύμφωνο. Ό,τι είπαν οι προλαλήσαντε συνάδελφοι επίση μου φαίνεται απόλυτα σωστό και Πράγματι, ότι προτείνουμε λιγότερο για πολύ περισσότερου δικαιούχου. Έχουμε και τη γεωγραφική εξάπλωση, αλλά και την αύξηση ε, ανθρώπων που είναι σε κατάσταση δύσκολη λόγω της κρίσης. Μειωμένοι πόροι για μεγαλύτερα προβλήματα. Εγώ θέλω να αναφέρω ένα πολύ συγκεκριμένο ζήτημα. Όπω γνωρίζετε, ε, εξαρτήσει για την επιστηστική βοήθεια προβλέπονται το Σεπτέμβριο και Οκτώβριο-Νοέμβριο είναι επιχειρησιακές για το επόμενο έτος. Οπότε γίνονται και οι αγορές και, τα αποθέματα. Όμως, με βάση τη συμφωνία, ο μηχανισμός προβλέπεται να λήξει στα τέλη του 2013. Και θέτω το εξή ερώτημα. Αν, όλος τυχαίως, δεν υπάρχει δημοσιονομικό πλαίσιο ή δημοσιονομική στήριξη για το συγκεκριμένο κανονισμό για το επόμενο Σεπτέμβριο. Τι θα γίνει, τι θα γίνει τότε. Θα έχουμε όχι απλά λιγότερους πόρους για περισσότερου δικαιούς, αλλά δεν θα έχουμε καν ε, πόρους, ούτε καν προοπτική για διάθεση κάποιων κονδυλίων. Αν λοιπόν το Σεπτέμβριο δεν έχει εγκριθεί ούτε το δημοσιονομικό πλαίσιο και δεν έχουμε προοπτικές για το 2014, θα είναι αδύνατον οι μη κυβερνικέ οργανώσει, οι οποίε συνήθω διαχειρίζονται αυτές, ε, αυτά τα θέματα, να διαχειριστούν την εξαρτήτη του 2014. Και εκεί θα έχουμε πραγματική καταστροφή. Γιατί είναι πάρα πολύ πιθανό να μην έχουμε σταθερέ μεσονομικέ προοπτικέ, να μην έχουν ψηφιστεί και υπό τι συνδίκε αυτέ είναι επίση πιθανό να μην έχουμε καμία λύση και για την επόμενη χρονιά, για του χρόνου. Διαρωτώ λοιπόν και θα κάνω και πρόταση πρώτες τροπολογία σχετικά. Διερωτώ λοιπόν μήπως θα μπορούσαμε να προβλέψουμε να ζητηθεί από το Ευρωπαϊκό Κεντρικό Ταμείο έστω προσωρινά να τροφοδοτήσει ε, με πόρους το Ταμείο αυτό για τους απόρους τουλάχιστον για αυτή την περίοδο. Ναι, ευχαριστώ πολύ. Κατανοώ το πρόβλημα. Το αντιλαμβάνομαι και εγώ. Και θα πρέπει να πιέσουμε και το Συμβούλιο να επιταχύνει έτσι ώστε μέχρι το Σεπτέμβριο να υπάρχει συμφωνία. Δεν είναι και ιδιαίτερα επίμαχο. Εντάξει, υπήρξαν κράτη-μέλη μεταξύ αυτών ε, το δικό μου κράτος που ήθελαν να το καταργήσουν τελείως το πρόγραμμα, αλλά τελικά εντάξει. Ε, ο Φρεντερίκ Νταρντέν και μετά ο Σουσέ Μανουέλ και οι υπόλοιποι. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Καταρχάς θέλω να ευχαριστήσω και εγώ τον εισηγητή Ντέρικ για, για το σχέδιο έκθεσης. Ως μέλος Επιτροπής Προπολογισμών και της Επιτροπής Απασχόλησης και ως συνεισηγητής για την πλατφόρμα αυτή, χαίρομαι που τελικά βλέπουμε να μονιμοποιείται αυτό το ταμείο για τους απόρους ε, και η πρικοδότησή του. Πράγματι έχει διευρυνθεί το πεδίο εφαρμογή, το εύρωσταλ, όπω είπαν και άλλοι συνάδελφοι, βλέπουν να μειώνονται οι πόροι. Και θα είναι σίγουρα ανεπαρκή για να καλυφθούν οι ανάγκε. Πιστεύω λοιπόν ότι θα πρέπει να παραμείνει προτεραιότητα προ την επιστηστική βοήθεια. Βλέπουμε ότι οι ανάγκε στι διαφορέ χώρε μέλη και ιδίω στο τοπικό επίπεδο αυξάνονται. Επίση, θα ήθελα να επιστήσω την προσοχή σα στον ορισμό ε, του κοινού στόχου δεν θα πρέπει να είμαστε περιοριστικοί ως προς τον ορισμό αυτό. Δύο-τρία ακόμη στοιχεία. Συγχρηματοδότηση. Προανέφεραν συνάδελφοι τα σχετικά. Νομίζω ότι πράγματι εδώ ελοχεύει ένα κίνδυνο και δεν θα πρέπει να τέθει τροχοπέδι με τον τρόπο αυτό στην χρησιμοποίηση του μελλοντικού ταμείου. Από την άλλη πλευρά όμω, αν υπάρχουν χώρε που θα επιθυμούσαν να συμπληρώσουν τον προπολογισμό, θα έπρεπε να υπήρχε αυτή η θελοντική βάση στη συγχρηματοδότηση. Να μην είναι δηλαδή υποχρεωτική, αλλά να είναι εθελοντική η βάση αυτή. Τέλος, δεν θα πρέπει να υπάρξει ε, ρήξη ε, της, ε, των παροχών. Από την 1η Ιανουαρίου 2014 θα πρέπει να μπορεί μέσω του Ευρωπαϊκού Ταμείου, δεν ξέρω εγώ ποιο άλλο ταμείο, να μπορεί να συνεχιστεί η βοήθεια, να μην υπάρξει διακοπή. Πρέπει έστω και προσωρινά να βρεθεί μια λύση. Ευχαριστώ. Ähm, ευχαριστώ. Έτσι κι αλλιώς το θέμα είναι ε, μήπως εμείς κάνουμε τέτοιες προσπάθειες για ένα πολύ καλό ε, πρόγραμμα, ένα πολύ καλό κανονισμό και να καταλήξουμε στα 2,5 εκατομμύρια, λέει η Πρόεδρος, που δεν είναι, είναι γελίο ποσό. Ε, Σας ευχαριστώ, Πρόεδρε. Και εγώ θα ήθελα να συγχαρώ τον εισηγητή διαγράφεται ευρεία συνένεση σε σχέση με την θέση του με βάση όλες τις ε, παρεμβάσεις ε, με τις οποίες συμφωνώ. Σε σχέση με τη στρατηγική Ευρώπη 2020 υπήρχε ένα στόχος που ήταν η μείωση του αριθμού των φτωχών στην Ευρωπαϊκή Ένωση και το πρόγραμμα αυτό σχετίζεται άμεσα με το στόχο αυτό. 20 εκατομμύρια φτωχοί φαίνεται να είναι ένα νούμερο παροχημένο. Σήμερα είμαστε πολύ πάνω από τα 20 εκατομμύρια φτωχούς και γι' αυτό θα έπρεπε να υπάρχει μεγαλύτερη ευελιξία όσον αφορά τα ποσά που κατευθύνονται στην επίτευξη αυτού του στόχου. Να είναι επαρκή όχι για τα 20 εκατομμύρια, αλλά για το πραγματικό αριθμό φτωχών που έχει αυξηθεί. Έχει αυξηθεί η φτώχεια γενικά στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Ε, το άλλο μου ερώτημα σχετίζεται δεν σχετίζεται άμεσα με αυτή την Επιτροπή. Πάντως αυτό το πρόγραμμα θέλει να αντικαταστήσει το πρόγραμμα επιστημιστικής βοήθεια που ήταν, δεν ήταν σε χρηματοδοτούμενο, ήταν 100%. Εδώ λοιπόν το ποσοστό συγχρηματοδότηση αυτό το νέο πρόγραμμα που έχει και διευρυμένο πλαίσιο να είναι και αυτό 100%. Στο προηγούμενο πρόγραμμα χρησιμοποιούνταν τα γεωργικά πλεονάσματα. Το ερώτημά μου λοιπόν είναι... Ε, τι έγινε, δεν έχουμε πια πλεονάσματα γεωργικά. Όχι. Τι γίνονται τώρα αυτά τα πλεονάσματα. Να θυμίσω ότι αυτό προκύπτει από μια απόφαση του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου που θα μπορούσαμε να τη χρησιμοποιήσουμε να χρησιμοποιήσουμε τα, πλεον, γεωργικά πλεονάσματα ε, όπου σε μια Ευρώπη που υποτίθεται ότι είναι αυτάρκης ε, είναι απαράδεκτο να μην εκμεταλλευτούμε τα γεωργικά αυτά πλεονάσματα και να πρέπει να έχουμε νομικές λύσεις για να μπορέσουμε να, να, να τα εκμεταλλευτούμε. Δεν ξέρω ακριβώς τον, αριθμό των πλεονασμάτων, ούτε ξέρω ακριβώς που πηγαίνουν αυτά αυτή τη στιγμή. Πάντως, εγώ συμφωνώ ε, με την έκθεση. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ πολύ. Ναι, όλα αυτά κανείς τα καταλαβαίνει που λέτε, αλλά είναι σαφές ότι έχουμε μια νέα πρόταση τώρα για το νέο πρόγραμμα, διότι το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο απεφάνθη ότι δεν είναι ε, υπόθεση της κοινή γεωργικής πολιτικής να βοηθάει τους ιδιαίτερα απόρους στην Ένωση και να τους δίνει επισυνδυστική βοήθεια. Αν τώρα εμεί έλθουμε και το προσθέσουμε αυτό, δεν ξέρω, ίσως χρειαστεί να ζητήσουμε από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να εκπονήσει νέα πρόταση για το τι θα γίνει με τα γεωργικά πλεονάσματα. Αλλά δεν μπορώ να φανταστώ τώρα η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και μάλιστα σε πολύ μικρό χρονικό διάστημα να είναι πρόθυμη να κάνει το παραμικρό. Γιατί από μόνοι μας δεν μπορούμε με δική μας πρωτοβουλία να κάνουμε την πρόταση αυτή. Γιώργεν, ευχαριστώ Γιώτα. Ευχαριστώ και τον εισηγητή για την εργασία του. Ε, μπορούμε να συμφωνήσουμε σε πολλά και εμείς. Απλώς θέλω να ρωτήσω κάτι για τους γεωργικούς πόρους. Έχει νόημα και μπορούμε να τεκμηριώσουμε μια τέτοια πρόταση, αλλά δεν ξέρω κατά πόσο ακολουθούν και τα χρήματα ε, από τον ένα τομέα έχουν μεταφερθεί στον άλλον κουνά στο κεφάλι σου. Δεν θα πρέπει όλα αυτά να μεταφορθούν γιατί ε, αλλιώ θα πρέπει να γίνουν περικοπέ σε άλλε θέσει του προπολογισμού του προγράμματο. Οπότε δεν λύνεται το πρόβλημά μα έρχεται να προσθεθεί και ένα καινούριο. Λέει και ο και επίσης γενικά είναι πολύ χαμηλό το ποσό στις χώρες κρίσης είναι πάρα πολύ δεινή η κατάσταση. Στην Ελλάδα είναι χειρότερη, αλλά και σε άλλες ισχύει. Έχει αυξηθεί η έδεια, έχουν αυξηθεί τα συσίτια και η τεχνική πλευρά επιμελητία χρειάζεται ενίσχυση. Και ε, το Συμβούλιο χαρακτηρίζεται από ένα κινησμό, πρέπει να πω, που έκανε τέτοια γενναία περικοπή στο συγκεκριμένο κονδύλι. Να το πούμε και αυτό. Και ένα τελευταίο για τη συγχρηματοδότηση, δεν μπορώ παρά να το υπογραμμίσω, από πλευράς μας συμφωνούμε με τον εισηγητή και επαυξάνουμε. Ευχαριστώ. Ja, vielen Dank. Äh, von Ευχαριστώ. Δεν είναι μεταφορά πιστώσεων, ε, γιατί είναι καινούριο του κουτιού εντός εισαγωγικών το πολιετές δημοσιονομικό πλαίσιο και το νέο πρόγραμμα αλλά δεν έχω την αίσθηση, την εντύπωση ότι είναι αρκετή η πρικοδότηση του προγράμματος. Ας σε πω, διαβάσεις και το κείμενο. Ε, είναι ένα υποπρόγραμμα του κοινωνικού ταμείου. Και ξέρουμε πού θα κατάληξει. Όταν κάτι είναι από την αρχή υποπρόγραμμα, τότε πολύ γρήγορα, όταν αυξηθούν οι ανάγκες, αντλούνται κονδύλια από το κοινωνικό ταμείο. Δηλαδή το παίρνουμε από τον ένα για να το δώσουμε στον άλλον. Είναι κάπως δύσκολα τα πράγματα. Τίποτα άλλο, ε, άλλος κανείς θέλει το λόγο, εισηγητής για να ολοκληρώσει. Yeah, yeah, Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Θέλω να ευχαριστήσω τους συναδέλφους για τις παρεμβάσεις τους. Νομίζω ότι όλοι εξέφρασαν την υποστήριξή τους και θα είναι χρήσιμα τα σχόλια. Αρχίζω με τον Γιάννη, θέλω να πω ότι συμφωνώ απόλυτα μαζί του και πράγματι οι κανόνες ε, για τα φιλανθρωπικά τρίματα και για τους Ο μικρό θα πρέπει να είναι όσο το πιο απλή και γι' αυτό ε, θα φροντίσω και εγώ. Και τα θετικά, τα τεχνικά ζητήματα που ανέφερε, προθεσμίες κτλ. θα τα λάβω υπόψη μου, είπε βέβαια θα καταθέσει και τις τροπολογίες του. Ο Τζιωβάνι είπε για την εξάπλωση ε, που τελικά σημαίνει ότι είναι πιο λεπτό το στρώμα, αν θέλετε, τη μαρμελάδα που απλώνουμε στη φέτα, άρα ε, λιγότερα χρήματα για τους περισσότερους δικαιούχους. Πράγματι, ε, έχουμε όλο και περισσότερα αισθήματα να καλύψουμε και παρανερχόμαστε στο θέμα της πρικοδότησης. Φτάνουμε στα 2,5 δις δηλαδή για την επταετία και αυτό είναι ένα πρόβλημα. Άλλοι συνάδελφοι ανέφεραν ε, τη συγχρηματοδοτηση τρει τέσσερι τουλάχιστον συνάδελφοι. Εγώ προσωπικά, όπου είναι δυνατόν, θα ήθελα να εξασφαλίσουμε το 100% χρηματοδότηση των ε, προγραμμάτων στα κράτη-μέλη. Παραλαμβάνω όμως έχουμε περικοπεί στο συνολικό ποσό και αυτό μας δημιουργεί προβλήματα. γιατί ίσως θα χρηματοδοτηθούν πολύ λιγότερα σχέδια, πολύ λιγότερα προγράμματα. Όλα αυτά βέβαια είναι θα είναι θέμα διαπραγμάτευσης και ίσως βρούμε κάποιους συμβιβασμούς. Ίσως έχουμε περισσότερη ευελιξία για τα νούμερα ή για τα συντελεστές συγχρηματοδότησης, τουλάχιστον για τα πιο φτωχά να μπορούν να εξασφαλίσουν τουλάχιστον αυτά το 100% της χρηματοδότησης και κάποια άλλα λιγότερα. Δεν λέω ότι είναι αυτή η άποψη. Ξέρω ότι είναι δύσκολη καιρή και πρέπει όλα να τα διαπραγματευτούμε στο μέλλον. Δεν θα πω κάτι περισσότερο. Να ευχαριστήσω τους συναδέλφους για μια ακόμη φορά. Ήταν καλή συζήτηση. Νομίζω ότι οι συνάδελφοι που μίλησαν ε, έδειξαν ότι με υποστηρίζουν και τους ευχαριστώ. Ja, vielen Dank. Ευχαριστώ πολύ. Προθεσμία κατάσταση τροπολογιών αύριο είπαμε στις 12 το μεσημέρι. Όσοι θέλετε να κάνετε τροπολογίες και θα ψηφίσουμε στις 26 Μαρτίου εμείς εδώ την γνωμοδότηση. Έτσι ώστε η Επιτροπή Επασχόλησης να την έχει εγκαίρως. Και ερχόμαστε στο σημείο 8 της ημερήσιας διάταξης ανταλλαγή απόψεων σχετικά με ενδεχόμενες περιπτώσεις του Ευρωπαϊκού Ταμείου κατά της παγκοσμιοποίησης. Είναι μια ιταλική περίπτωση αυτή. Θα μας την εξηγήσει ο Φρεντερίκ Νταρντέν. Ist Σας ευχαριστώ. Θα είμαι σχετικά σύντομος. Θα ήθελα να σας πω ότι πρόκειται για 1.517 εργαζόμενες, εργαζόμενους στις καικές συσκευές, 700... 7.750.000 ε, ευρώ και προτείνω στην έκθεσή μου να χορηγηθεί η ενίσχυση. Ξέρω πως υπάρχουν τροπολογίες που έχουν κατατεθεί από την Επιτροπή Απασχόλησης και που θα πρέπει να έρθουν τις επόμενες μέρες. Ένα, ένα που χρειάζεται την υποστήριξή σας. Gibt es von den Kollegen oder eine Kollegin? Δεν ξέρω, υπάρχουν συνάδελφοι που θέλουν το λόγο για αυτό το θέμα. Κανείς. Ωραία. Τροπολογίες. Μπορείτε να καταθέσετε για αυτό το θέμα. Μέχρι αύριο, τις 12 το μεσημέρι επίση. Για να ψηφίσουμε στις 20 και 21 του μηνός Μαρτίου εδώ στην Επιτροπή μας. Μάλλον στις 20. Γιατί στις 20 ψηφίζει και η Επιτροπή Απασχόλησης για να προκάνει. Ωραία. Ερχόμαστε στη μία 15 της ημερήσιας ε, διάταξης, πολιτική ακινήτων. Keine, keine... Δεν έχουμε νέα τίποτα ε, επίκαιρα ζητήματα προς ενημέρωση για τα ακίνητα, αλλά μας λείπει η Αν Γένζεν. Χάσαμε την εισηγήτριά μας στη Γενική για τον προπολογισμό του 2014. Οπότε να ρωτήσουμε τους ε, εισηγητές για το προϋπολογισμό του Κοινοβουλίου. Ε, η Μόνικα για το 6, αγαπητή πρόεδρε η κυρία Χολμάγερ, δεν έχουμε τίποτα τόσο το καινούριο ε, Σήμερα την Παρασκευή έστειλα στους συναδέλφους ένα πρώτο προσχέδιο ε, της έκθεσης για την κατάσταση προβλέψεων του Κοινοβουλίου ε, και σας αναφέρω τα κυριότερα σημεία ε, από την κοινή ομάδα εργασίας, τα μέτρα ας πούμε οικονομίας που έχουμε λάβει ήδη και άλλες διαρθρωτικές αλλαγές, καθώς επίσης και αυτά που μας παρουσίασε εδώ Γενικό Γραμματέας του Κοινοβουλίου. Αν θέλετε να τα κοιτάξετε, με την ησυχία μας να τα συζητήσουμε, δεν έχουν ληφθεί καθόλου προ... καταρτικές αποφάσεις. Ε, στα πλαίσια της έκθεσης ε, θα πρέπει να πούμε ότι είμαστε υπέρ και νέων διαρθρωτικών αλλαγών για να ε, βελτιωθεί ε, η υποστήριξη του έργου των βουλευτών και επίσης ε, να έχουμε πιο ισχυρή εκτίμηση των επιπτώσεων που έχει η νομοθεσία και όταν ψηφίζουμε για νέες οδηγίες ή νέους κανονισμούς θα πρέπει να έχουμε τη σωστή επικούρηση από εμπειρογνώμονες όσο και ειδικού στο εσωτερικό του Κοινοβουλίου. Γνωρίζετε ήδη ότι Έχουμε ένα ιδιαίτερο προϋπολογισμό φέτος. Γιατί, γιατί η τελευταία χρονιά της θητείας, το 2014, με συνέπεια την εξή. Από όσα μας έχει πει μέχρι τώρα η διοίκηση του Κοινοβουλίου, μόνο 2,20% των δαπανών αφορά, η αύξηση δηλαδή αφορά αποκλειστικά ε, το τέλος της θητείας. Γιατί έχουμε εκλογές, γιατί οι συνάδελφοι φεύγουν, ε, άρα υπάρχει και κάποια οικονομική επιβάρυνση και νομικές ε, υποχρεώσεις του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου για συνέχιση της χρηματοδότησης των πρώην βουλευτών και μετά έχουμε και νέες υποχρεώσεις για τη χρηματοδότηση για τις απολαβές των νέων βουλευτών. Επίσης μας είπαν ότι ε, στον κανονικό προϋπολογισμό, δηλαδή όχι σε περίοδο εκλογών, εγώ θα επιθυμούσα πάρα πολύ να παραμείνουμε κάτω του ε, πληθωρισμού και τώρα το Προεδρείο προτείνει για τον τομέα αυτό που αφορά την αύξηση των απολαβών των ε, υπαλλήλων, διαρθωτικών αλλαγών και άλλων θέσεων και τίτλων του προϋπολογισμού. Δεν θα ακολουθήσουμε το τιμάριθμο 1,92% που είναι πληθωρισμός αλλά θα περιστούμε στο 1,3%. Αλλιώς θα ξεφύγει πολλή αύξηση ε, ακριβώ ε, και λόγω της ε, αλλαγής της θητείας. Επίσης 13,6 εκατομμύρια μόνο που θα μας κοστίσει η Κροατία που για πρώτη φορά είναι πλήρης έτος πλήρες το στον προπολογισμό και το κόστος που επιφέρει η ένταξη της Κροατίας και κάτι άλλο Όταν ε, αποφασιστεί και αν ένας νέος κανονισμός υπηρεσιακής κατάστασης, που διέπει δηλαδή τους υπαλλήλους, θα πρέπει το Προεδρείο αντίστοιχα να δράσει. Δηλαδή έτσι θα προκύψουν κάποιες αλλαγές και μάλλον και ε, ουσιαστικές οικονομίες αυτή τη στιγμή ολοκληρωθούν οι διαπραγματεύσεις και οι συζητήσεις. Και θα δούμε λοιπόν ανάλογα με τις αλλαγές, θα έχουμε ένα πολύ συγκεκριμένο δικό χάρτη, να φύλλο για να δούμε πώς όλα αυτά θα εφαρμοστούν στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Αυτό αφορά τη συνταξιοδότηση, ζητήματα εβδομαδιαίου ωραρίου, ε, ταξίδια και τα λοιπά άδειες, Αυτά τα συζητάει η κυρία Ροτ Μπέρεντ και ο νέος λοιπόν κανονισμός θα ισχύσει και οι κανόνες θα αφορούν τους ενδιαφερομένους. Επίσης το 2009 είχαμε ένα προπολογισμό ε, που ήταν η προηγούμενη ε, λήξη της θητείας και μπορούμε να το συγκρίνουμε με το 2014, η αύξηση ήταν ουσιαστικά πάνω από το 5%. Τώρα έχουν αλλάξει τα πράγματα γιατί σε καιρούς κρίση πρέπει να είναι κανείς πιο προσεκτικός στη διαχείριση των οικονομικών. Αλλά αυτό το μεταβατικό κόστος δεν μπορούμε να το αποφύγουμε. Αύριο στη συνδιαλλαγή, αν συμφωνήσουν και οι συνάδελφοι, με χαρά να κάνω κάποια ερώτηση για αυτό το μεταβατικό κόστος. Πάντως είμαστε υποχρεωμένοι ε, δια νόμου να καλύψουμε κάποιες δαπάνες όταν αλλάζει η θητεία, φεύγουν βουλευτές, έρχονται νέοι. Ε, έχουμε επιπλέον οικονομική επιβάρυνση και δεν μπορούμε να τα αλλάξουμε αυτά. Ε, Επίση, χαίρομαι που αύριο θα πάμε στην προ-συνδιαλλαγή και με την κοινή ομάδα δράσης ομάδα εργασία μάλλον του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Θα συζητήσουμε αυτά τα θέματα μέχρι το φθινόπωρο Θέματα τα οποία παρουσίασε ήδη τουλάχιστον μια φορά στην Επιτροπή μας ο Γενικός Γραμματέας με τους αρμόδιους αντιπροέδρους. Και να πω και κάτι ακόμα. Το κτίριο ΚΑΔ στο Λουξεμβούργο το παρακολουθούμε πάρα πολύ στενά. Πρέπει να σας πω ότι από ό,τι φαίνεται ο δεύτερος διαγωνισμός ε, είναι μεγάλη επιτυχία και μεγάλη οικονομία θα μείνουμε κάτω του προπολογισμού που είχαμε προβλέψει και ε, μπορούμε επίσης να εξοικονομήσουμε πολλά χρήματα. Οπότε η κοινή μας γραμμή που την τηρήσαμε έτσι με πείσμα πρέπει να πω και με στένος στέφθηκε με επιτυχία. Έχει κάπως συμμαζευτεί το κόστος, είναι λογικό και δεν θα ζήσουμε μεγάλες ε, εκπλήξεις, ε, αλλά θα είναι χαρμόσυνο αυτό το γεγονός μετά τον πρώτο άγωνο διαγωνισμό ναι, σε ό,τι αφορά τον προπολογισμό του Κοινοβουλίου, θεωρώ και εγώ θα πρέπει να καταγράψουμε πρώτα όλε μα τι επιτυχίες, πριν βγούμε πάλι και λέμε ότι χρειάζονται περισσότερες οικονομίε. Εν πάση περιπτώσει, ο George Λάιον και μετά η ε, Edith Χέρτσοκ. Ε, Ευχαριστώ. Θέλω να ευχαριστήσω και τη Μόνικα για την ενημέρωση αυτή. Για ένα πολύ σημαντικό θέμα. Πρώτα απ' όλα, σε ό,τι αφορά το κτίριο ΚΑΤ, ε, είχαμε κάποιες εξελίξεις. Το, ε, για, με τους διαγωνισμούς είχαμε κάποιες προσφορές 30% πιο πάνω και κάποιες 10% κάτω. Σε ό,τι αφορά τώρα το συνολικό προϋπολογισμό, Καταλαβαίνω ότι πρέπει αυτό το κόστος λόγω των ευρωεκλογών να, το απορροφήσουμε, αλλά πιστεύω ότι θα πρέπει να φροντίσουμε οι προτάσεις που ενέκρινε το Προεδρείο να φροντίσουμε το 2013 να μην έχουμε αύξηση πάνω από το επίπεδο του προπολογισμού. Εμεί προσπαθούμε να αλχιστοποιήσουμε ω Κοινοβούλιο την αυξήση αυτή, αλλά ω Επιτροπή νομίζω προπολογισμού πρέπει να πιέσουμε ακόμη περισσότερο. Θα είναι πάρα πολύ δύσκολο να είναι πολύ πάνω από τον πληθωρισμό αυτό το ποσό σε έτος ε, προεκλογών. Είναι ένα άπαξ, άπαξ ποσό. Θα έπρεπε να προσπαθήσουμε, πιστεύω, να τι μειώσουμε ακόμη περισσότερο αύριο ίσως με το Προεδρείο θα μπορούσαμε και με το Γενικό Γραμματέα να αρχίσουμε ήδη να διερευνούμε τις σχετικές πιθανότητες. Ευχαριστώ, η Edit. Ε, ε, ε, I Ευχαριστώ, Πρόεδρε με χαρά θα σας πω τι έγινε στην ομάδα. Καταρχήν θα ήθελα να ζητήσω από τον γραμματέα της Επιτροπής να σέβεται καλύτερα το χρόνο για να μπορούμε να προετοιμαστούμε καλύτερα. Οι εκτιμήσεις ήρθαν σήμερα το πρωί στις 10 το πρωί σήμερα ε, και είχαμε πολύ λίγο χρόνο να τα εξετάσουμε. Ίσως λοιπόν θα πρέπει να ξαναδούμε την διαδικασία μας. Βλέπω ότι υπάρχουν δυσκολίες και ότι είναι περίπλοκα τα θέματα. Ξέρω πως η απόφαση του Προεδρείου δεν έχει υπάρξει ακόμα αλλά αν θέλουμε να έχουμε ασφαλή πλειοψηφία εδώ, θα πρέπει να ανταποκρινόμαστε στις μίνιμουμ ανάγκες των μελών. Να πω επίσης εδώ ότι αυτοί που προετοιμάζουν τις, ε, τις καταστάσεις προβλέψεων είναι τα καλά παιδιά, ενώ εμείς που είμαστε εδώ είμαστε τα κακά παιδιά. Δεν μπορεί να είναι πάντα έτσι η διοίκηση να είναι τα καλά παιδιά και εμείς να είμαστε υπεύθυνοι για όλες τις ε, ε, περικοπές. Εδώ τώρα υπάρχουν διάφορα καλά στοιχεία. Ε, θα το σκεφτούμε για να υποβάλουμε τροπολογίες. Το 3,48% φαίνεται να είναι πολύ ψηλό, περιβολικά ψηλό και πολύ δύσκολο να το εξηγήσουμε. Γι' αυτό χρειάζεται καλή καλύτερη αιτιολόγηση για κάποια από τα κεφάλαια και Πιστεύω ότι αυτό είναι πολύ σημαντικό, όπως επίσης είναι πολύ σημαντικό να δούμε πού μπορούν να γίνουν περαιτέρω εξοικονομήσεις. Οποιαδήποτε συμβουλή από τη διοίκηση, από συναδέλφους, είναι ευπρόσδεκτη. Θα ήθελα λοιπόν να πω ότι στο σχέδιο έκθεσης Θεωρούμε πως η συγγήτρια προχωρά λίγο περισσότερο από τα συνεχιζόμενα προγράμματα στην ομάδα εργασία. Εμείς διαφωνούμε λοιπόν σε αυτό το στάδιο να πάμε στο λεπτομερές κείμενο στην έκθεση για τον προπολογισμό, γιατί η ομάδα εργασία είναι υπό εξέλιξη. Από την άλλη πλευρά όμως, Οι προτάσεις θα πρέπει να είναι έτοιμε εγκαίρω να μπουν μέσα στην έκθεση. Συμφωνώ και με τον προηγούμενο μιλητή ότι για την κτηριακή πολιτική υπάρχει αύξηση 18,3 ε, αύξηση που είναι η μεγαλύτερη αύξηση πέρα από τα μεταβατικά κόστη για την εκλογική χρονιά Θέλουμε να βάλουμε λοιπόν στο κείμενο ότι οι εξοικονομήσει δεν επιτέθηκε από τη διοίκηση, αλλά από το, μετά από αίτημα της, δημοσιονομικής, της Επιτροπής Προπολογισμού. Και είναι πάρα πολύ σημαντικό να αναφέρουμε πως ε, εμείς εδώ και τα μέλη της Επιτροπής μας στην Ολομέλεια άσκησαν πίεση για τη δεύτερη, το δεύτερο διαχωνισμό. Τελευταία δήλωση. Νομίζω πως όλοι συμφωνούμε ότι τα χρήματα που πρέπει να πληρωθούν κατά τη μεταβατική περίοδο για εκείνα τα μέλη και για εκείνα στις υπαλλήλους που φεύγουν από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο στο δεύτερο ήμιση του έτους θα πρέπει να πληρωθούν. Αλλά εδώ νομίζω πως χρειάζεται λίγο, λίγο περισσότερες λεπτομέρειες για το πόσα χρήματα πληρώθηκαν το 2009 από τα κράτη-μέλη στην προηγούμενη εκλογική χρονιά. Η αύξηση αυτή να είναι αύξηση στο επίπεδο Ένωση, αλλά όχι πραγματική αύξηση που πληρώθηκε από τα κράτη-μέλη. Γιατί η μισθοί και τα επιπλέον κόστη πληρώθηκαν από τα κράτη-μέλη στις προηγούμενες εκλογές. Έχουμε μια αναπόφευκτη αύξηση λοιπόν και ίσως θα μπορούσαμε να αποφασίσουμε το 2009 να ε, αντλήσουμε από το αποθεματικό. Και ίσως θα πρέπει να ξαναδούμε την διαδικασία γιατί είναι πάρα πολύ δύσκολο να απορροφηθούν όλα αυτά σε ένα χρόνο. Τώρα όμως πρέπει να, δούμε, να ανταποκριθούμε στην κατάσταση αυτή και το Κοινοβούλιο θέλει να αποτελέσει πρότυπο καλού εργοδότη. Σας ευχαριστώ πολύ. Αυτά είναι τα βασικά που ήθελα να πω εξ ονόματος των σοσιαλιστών. Ja, vielen Dank. sonst noch Wortmeldungen? Ευχαριστώ. Θέλει άλλος κανείς να μιλήσει. Α, έχουμε και άλλο εισηγητή. Ναι. Η εισηγήτριά μας για τον προπολογισμό του 2014 όμως αποσιάζει. Και μόλις τελειώσουμε αυτό το σημείο, ε, θέλω να ρωτήσω τους εισηγητές για το πολιτές δημοσιονομικό πλαίσιο και ελπίζουμε να έρθει η κυρία Γέντσεν μέχρι τότε. Ε, Μόνικα, θες να ολοκληρώσει εσύ, Χολμάγερ. Ευχαριστώ πολύ, κυρία Πρόεδρε. Θα ήθελα να ξαναφέρω λίγο τα στοιχεία για να καταλάβουμε περί τίνος πρόκειται. Τι συμβαίνει τώρα. Αν δούμε τη σύγκριση με το περασμένο έτος, για τον προπολογισμό αυτό καθ' αυτό, αφήστε το κόστος που προκύπτει από τη λήξη της θητείας, θα είμαστε κάτω από το επίπεδο του 2013. Στις θέσεις του προπολογισμού, μάλιστα, υπάρχουν και αρνητικά πρόσωπα, δηλαδή μειώσεις. Καθόλου αύξηση. Ε, μετατοπίσεις μόνο εντός των κονδυλίων, παράδειγμα, προς την επιστημονική υπηρεσία και ε, στην πολιτική ακινήτων ε, υπάρχει μετατόπιση διότι έχουμε τώρα εξαγοράσει τα κτίρια και έχουμε κόστος βέβαια για τη συντήρηση των κτιρίων μας, αλλά ε, μειώνονται σημαντικά τα μισθώματα και το leasing που πληρώναμε. Λοιπόν, υπάρχει μετατόπιση από ε, μια γραμμή προπολογισμού σε μια άλλη. Και κάτι άλλο που θα πρέπει αύριο να δούμε από κοινού είναι αυτό το μεταβατικό κόστος και ποια είναι η διαφορά σε σχέση με το 2009. Ότι δεν πληρώνουν πια τα εθνικά κοινοβούλια, Bundestag ή η αυστριακη Βουλή και η Ολλανδία για τους Ολλανδούς, αλλά για πρώτη φορά ε, ε, το κοινοβούλιο επομίζεται το κόστος. Για έχουμε και δικαίω κατά την άποψή μου εγκρίνει ε, το καθεστώς των βουλευτών και ερχόμαστε τώρα να βρούμε τις συνέπειες μπροστά μας. Έχουμε γίνει επιτέλους κανονικό κοινοβούλιο για να το πω έτσι. Δεν είμαστε ένα κοινοβούλιο που βασίζεται ε, στις υπηρεσίες των Εθνικών Κοινοβουλίων, αλλά ε, καλύπτει τις δαπάνες του από το καθεστώς των βουλευτών σε μεγάλο βαθμό το ίδιο. Ε, αυτό αποφασίσαμε, τώρα θα πρέπει να βάλουμε και το χέρι στην τσέπη. Και το Προεδρείο το αποφασίζει αυτά. Κάτι που θα θεωρούσα δυσάρεστο είναι να βρούμε διάφορα κόστη μπροστά μας που για λαϊκιστικούς και μόνο λόγους δεν τα έχουμε γράψει στον προπολογισμό. Αφού υπάρχουν μεταβατικά κονδύλια, είμαστε υποχρεωμένοι να τα καλύψουμε, τα καλύψουμε όπως έκανε και κάνει άλλωστε κάθε εθνικό κοινοβούλιο και δεν τον φυσβητεί κανείς. Ευχαριστώ την Edith Herzog που έθεσε αυτά ε, τα ζητήματα, θα τα ρωτήσω τι γίνεται με τις μεταβατικές ρυθμίσεις και με βάση ε, ποιων ε, αριθμών έχουν υπολογιστεί αυτά τα ποσά. Είναι ρεαλιστικά, είναι ε, έτσι γενναιόδωρα υπολογισμένα και δεν μπορούμε να τα αλλάξουμε με αλλαγή των θέσεων του προϋπολογισμού και συμφωνήσαμε το Κοινοβούλιο να κοινοποιήσει την ε, ημερομηνία των εκλογών και να υπάρχει συμμετοχή ε, όχι 30 και 40% να ξέρει ο κόσμος πότε γίνονται οι ευρωεκλογέ και να είναι ενημερωμένοι. Δηλαδή και να ενημερώνει το Κοινοβούλιο για αυτά. Να είμαστε μεν ε, ε, φιδωλοί στη διαχείριση και οικονόμη, αλλά ε, δεν θα πρέπει να επιλέγουμε αλακάρτ γραμμές του προϋπολογισμού, αλλά ε, η μόνη δυνατότητα να γίνει αυτό, το είδαμε και την περασμένη φορά, είναι με ε, διαρθρωτικές αλλαγές. Τώρα κόβεις λίγο δεξιά και αριστερά, δεν βοηθάει πραγματικά, δεν λειτουργεί. Δεν υπάρχουν αυξήσεις στον προϋπολογισμό. Οι αυξήσεις των μισθών των υπαλλήλων θα πρέπει να ληφθούν υπόψη. Δεν μπορούμε να τις αγνοήσουμε απλούστατα. 1,3% είναι ένας προσεκτικός προϋπολογισμός και συγκρατημένος και το 2009 ε, την περασμένη φορά που άλλαξε το κοινοβούλιο το κόστος ήταν 5,33% και δεν είχαμε και ένταξη νέου κράτους για να επομιστούμε επιπλέον δαπάνες. Δηλαδή το 2014 είναι όντως ξεχωριστή χρονιά, χρειάζεται προσοχή, σύνεση αλλά να μην περιορίσουμε και τις δυνατότητες ε, δράσης και λειτουργίας μας, ούτε το 2014, να τις διατηρήσουμε. Ευχαριστώ πολύ. Θα τα ξαναπούμε αυτά τα θέματα επανειλημμένα, όχι μία φορά μόνο. Αύριο ε, είναι η πρώτη αυτή προκαταρκτική συνεδρίαση, το μεσημέρι 2 με, 12 ε, με 2, συγγνώμη. Και θα δούμε πώς θα προχωρήσουμε. Το Προεδρείο πότε αποφασίζει για αυτά τα θέματα. Τη Δευτέρα, την άλλη εβδομάδα ήδη. Έπρεπε να είχαν αποφασίσει την περασμένη εβδομάδα. Αλλά η κατάσταση προβλέψεων ήρθε πάρα πολύ αργά ακριβώ γιατί δεν αποφάσισε το Προεδρείο. Εξού και η όλη καθυστέρηση στην κατάσταση προβλέψεων. Τώρα προβλέπουν Α, στις 11 του μηνός λέει, δεν έχει αλλάξει. 11 Μαρτίου προθεσμία κατάσταση τροπολογιών. Στις 11 Μαρτίου θα αποφασίσουν και τότε λύγει και η δική μας προθεσμία για την κατάσταση τροπολογιών, 11 Μαρτίου. Μάλιστα και από εκεί και πέρα βλέποντας και κάνοντας. Συμφωνείς με αυτά τα χρονοδιαγράμματα ή μπορούμε να αναβάλουμε την προθεσμία για την κατάθεση τροπολογιών, να την παρατείνουμε. Αν δεν διαμαρτυρηθούν τα πλήθη μπορούμε να την αλλάξουμε. Λοιπόν, 12 Μαρτίου στις 3 η ώρα το μεσημέρι λίγη προθεσμία τότε για τις ε, τροπολογίες, για να ξέρουμε τι θα αποφασίσει το Προεδρείο και αντίστοιχα να δράσουμε. Θα τα πω και στην Έντιτ και στη Χάνα που δεν μ' ακούνε. Η προθεσμία για την κατάθεση τροπολογιών τώρα άλλαξε, έχει 11 Μαρτίου, 12 του μηνός. Εντάξει, λέει η κυρία Ωραία. Τώρα κανονικά θα έπρεπε να συζητήσουμε τον προπολογισμό της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για το 2014. Η Αν Γένσεν κολλείεται, είναι σε άλλη επιτροπή και πρέπει να μιλήσει για αυτά τα θέματα εκεί. Αλλά εκκρεμεί ακόμα το σημείο 4 στη μέση διάταξή μου. Το πολιτές δημοσιονομικό πλαίσιο. Την περασμένη φορά μακρηγορήσαμε λίγο περισσότερο. Παρ' όλα αυτά θα ήθελα να ζητήσω από τους ε, εισηγητές να μας πούν αν πρέπει ε, να μας πούν σήμερα τίποτα καινούριο, υπάρχει τίποτα πιο πρόσφατο, πιο ε, νέο. Να αρχίσουμε από τον Ιβάιλο Κάλφιν η αλλαγή. Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε. Δεν έχουμε και τίποτα το τόσο καινούριο με τον Ράιμερ. Επεξεργαζόμαστε ένα σχέδιο ψηφίσματος για το Κοινοβούλιο Είχαμε κάποιες πρώτες αντιδράσεις και τώρα προσπαθούμε να οριστικοποιήσουμε το κύμα των διασυγητών και ελπίζω αύριο να μπορέσουμε να το διανύμουμε στις πολιτικές ομάδες για να έχουν τις διαβουλεύσεις τους. Αυτό όμως το στάδιο δεν έχω να προσθέσω κάτι παραπάνω. Καλώς. Δεν έχεις τίποτα να προσθέσεις παραπάνω. Ωραία. Μήπως έχει Κανένα άλλο. Όχι. Δεν έχετε τίποτα άλλο να συζητήσουμε γιατί έχουμε πρόβλημα. Πείτε κανένα θέμα. Wir wollten, Κανονικά θέλαμε να συζητήσουμε με την Αν Γένσεν για την διαπραγματευτική εντολή για τον τριμερή διάλογο, αλλά δεν είναι εδώ η κυρία Γένσεν. Λοιπόν, δεν θέλω να σας κρατήσω με το ζόρι. Το έχουμε συζητήσει την περασμένη Πέμπτη. Ξέρουμε έτσι και λιώς περί τίνος πρόκειται και η ίδια η Αν Γέννησεν τα ξέρει αυτά τα θέματα. Την άλλη εβδομάδα, τη Δευτέρα, συνεδριάζουν ξανά οι συντονιστές. Λοιπόν, καλό σας υπόλοιπο Δευτέρας και τα ξαναλέμε την άλλη Δευτέρα. Χαίρετε.